Καλό καθίστε σε μισό λεπτό θα ξεκινήσει η συνεδρία σας. Otwieram posiedzenie. Κυρίσω την ε, έναρξη της ε, συνόδου, περίοδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπή 28 του 2009. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να πω δύο λόγια. Όπως γνωρίζετε, πριν από δέκα ημέρες, ο Λέχ Κασίνσκι, πρόεδρος της Πολωνίας, ε, κύρωσε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και μάλλον πέρα από τι συνθήκε Λισαβόνα και έχουμε θυσιάσει